Ευχαριστώ την Επιτροπή, ευχαριστώ όλους για την κατανόησή τους αλλά επίσης για τη συνεργασία τους. Τέλειωσε η συζήτηση και η ψηφοφορία είναι αύριο το μεσημέρι. Πριν προχωρήσουμε στο χώρο των ερωτήσεων, ε, έχουμε ε, αλλαγές αντιπροσωπείες των σοσιαλιστών ο κύριος γίνεται ε, πλήρες μέρος στην EEA και ο κύριος Βάισεν στην ε, ε, ε, αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης. Ε, ζητώ συγγνώμη από ε, την Επιτροπή και από το Συμβούλιο διότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτήν τη διαδικασία. Συνήθως εναλλάσσω με την κυρία Γουόλης. Η πρώτη ερώτηση παριθμών 1 είναι από τον κύριο Πόσελτ σχετικά με το κράτος δικαίου στη Σερβία. Ε, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου ήταν έτοιμη. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ουγγρικά αν μου το επιτρέπετε για να απαντήσω στην ερώτηση σχετικά με τον, το κράτος δικαίου στη Σερβία ε, ε, ε, στην απόφαση του Συμβουλίου του περασμένου έτους το Συμβούλιο είπε ότι εξήτασε την κατάσταση και ε, έχει ε, δημοσιεύσει τα απορίσματα λέγοντας ότι η Σερβία συνεχίζει να συμμορφώνεται στις διατάξεις σταθεροποιήσεως που προβλέπει η Συμφωνία Συνδέσεως αλλά θα πρέπει να βελτιώσει την δημόσια διοίκηση, τις δικαστικές αρχές, να καθιδρύσει το κράτος δικαίου και να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις δεν συζητήσαμε το κράτος δικαίου στη Σερβία στο Συμβούλιο για τη συγκεκριμένη περίπτωση την οποία μας υποβάλλει ο ερωτών. Κύριε Πόσελ, θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, ε, όταν ε, έκανα την ερώτηση υπήρχε ε, μία δίκη ε, μίας ομάδος υπηκών προελεύσεως Αλβανικής που έλαβαν την ανώτατη πηγή, δεν θα, ε, ανώτατη ποινή. Δεν θα έπρεπε όμως να έχει υπάρξει ε, ένας έλεγχος και θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε τη συγκεκριμένη περίπτωση την, επί της οποίας έκανα την ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο σχετικά με οποιοδήποτε θέμα είτε πρόκειται για τη διεύρυνση είτε για τις ε, συμφωνίες συνδέσεως πρέπει να παρακολουθεί ε, από το 1993 τα κριτήρια τα οποία είχαν καταρτιστεί και τα οποία πρέπει να, εφαρμόζονται. Δεν έχουμε λοιπόν άλλο τρόπο παρά να παρακολουθούμε αυτά τα κριτήρια κατά τις διαπραγματεύσεις. Βέβαια σημειώνω την ερώτησή σας και ε, η Ουγγρική Προεδρία θα ερευνήσει το πρόβλημα και όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις διαδικασίες έτσι και για την Σερβία θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα. Να προχωρήσουμε στο δεύτερο θέμα από τον κύριο Χίγκινς, Ο κύριος Κασπάρη διαδικαστικό. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω και μία δεύτερη ερώτηση η οποία ακολουθεί την ερώτηση του κυρίου Πόσελτ γιατί ε, ρώτησε ο κύριος Πόσελτ ε, πώς, τι θα γίνει σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση ε, προς το Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να έρθει το Συμβούλιο σε επαφή και η Προεδρία με τις υπεύθυνες αρχές στην αυτή δεν ήταν μία διαδικασία μπλε ε, κάρτας. Κανονικά θα έπρεπε να έχετε ε, ζητήσει ε, το, να εγγραφείτε από τη γραμματεία. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, θα λάβουμε υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο και το πνεύμα με το οποίο εξετάζει το Συμβούλιο τέτοιε υποθέσει. Μπορώ να σας πω ότι οι διαδικασίε είναι υπό εξέλιξη. Υπάρχει μια νέα φάση των διαπραγματεύσεων. Η Σερβία έχει απαντήσει στο ερωτηματολόγιο που κατέθεσε η Κομισιόν στις 21 ε, Ιανουαρίου η Σερβία μας έδωσε τις απαντήσεις της ε, και βέβαια κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων κάθε σημαντικό θέμα θα πρέπει να μελετηθεί από πλευρά της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στη δεύτερη ερώτηση του κυρίου Χίγκιν για τις μικρομεσαίες και την Ουγγρική Προεδρία. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν ζωτικό ρόλο στις ευρωπαϊκές οικονομίες για να βελτιωθούν οι κανονισμοί πλαίσιο είναι μία από τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας. Στους επερχόμενους μήνες η Προεδρία θα επιστιάσει την προσοχή της στην στρατηγική 2020 και τις ε, πρωτοβουλίες φλέξη για τις βιομηχανικές πολιτικές και την καινοτομία για ε, την εφαρμογή αυτών και την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μόνο το 8% των, των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων ε, κάνουν ε, διαμεθοριακές δραστηριότητες. Η έκθεση του Μάριο Μόντι επίσης ε, τονίζει πως για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ε, ιστορικής αγοράς θα πρέπει να εξαλειφθούν όλα τα εσωτερικά εμπόδια και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω οδηγιών και κυρίως τις, τις οδηγίες περί υπηρεσιών που έχει συζητηθεί επί μακρόν με τη σωστή της και ταχεία ε, εφαρμογή της. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με τις πληρωμές και τις διαμεθοριακές δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολύνονται από τα σχετικά φορολογικά καθεστώτα και θα πρέπει να υπάρχει και ευρωπαϊκό καθεστώς βρεσιτεχνιών για να ευνοηθούν οι μικρομεσαίες και το Κοινοβούλιο την Τρίτη έλαβε μια πολύ θετική απόφαση ως προς αυτό το θέμα, δηλαδή το θέμα του, των ευρεσιτεχνιών. Να ενθαρρυνθούν επίσης οι ΜΜΕ για να ε, συμμετέχουν σε καινοτόμες επενδύσεις. Επιπλέον θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην πράξη για τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αναθεώρηση αυτής. Θα θέλαμε να εφαρμόζουμε μια καθολική προσέγγιση στη νέα βιομηχανική, ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική μας και να εντοπίσουμε όλους τους φραγμούς κάθε τύπου που εμποδίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε αυτές να αποτελέσουν τραχοκοκαλιά της πράσινης οικονομίας. Επιπλέον, είναι στόχος μας να εισάγουμε πιο μοντέρνους κανονισμούς που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ. Θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε τις δυνατότητες ε, λειτουργίας των... και κίνησης των ε, ΜΜΕ. Να σας θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε πολύ σημαντικές αποφάσεις 4 Φεβρουαρίου να αφορά την κοινοτομία και ένα από τα βασικά ζητήματα για το πώς ε, μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να σας πω ότι είμαστε πεπισμένοι και δεσμευμένοι ώστε τα κοινοτικά μέσα αλλά και πλονεκτικά και όροι πίστοση να δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια. Τέλος, να προσθέσω ότι η Προεδρία μας θα καταθέσει προτάσεις στο Συμβούλιο για πολιετή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και για την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση αυτών των προγραμμάτων που θα συμπεριλαμβάνουν πολύ συγκεκριμένα μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως για ο μηχανισμός ε, κατανομής του κινδύνου. Κύριε Higgins, για επερώτηση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία που βρίσκεται εκεί που βρίσκεται σήμερα και καλωσορίζω τα όσα μας είπε η υπουργό. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η γραφειοκρατία. Και ο πρόεδρος Μπαρόσο είπε το 2004 ότι θα έκανε κάτι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπιστεί αυτή τη δυσκολία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Όταν λοιπόν ακούμε τα όσα μας είπε η Ουγγρική Προεδρία, θα πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ευτυχής και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό γιατί προκαλεί πολλές δυσκολίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριο Μπαλσίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ, αγαπητή Υπουργέ, το 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε ένα πακέτο 50 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα έπρεπε να εξυπηρετήσει τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι εκθέσει όμως που έχουμε μέχρι στιγμή είναι ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αρκετά αυτά τα χρήματα και κυρίως χρησιμοποιήθηκαν από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ωστόσο δεν επωφελήθηκαν σε επαρκή, επαρκές επίπεδο. Πώς λοιπόν εσείς θα προωθήσετε την χρήση τέτοιων κονδυλίων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Uh, Η κυρία Σίνκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι συμφωνούν. Νομίζω ότι συμφωνούν. Είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι μία γραπτή δήλωση την οποία στηρίζει ο Μάλκομ Χάρμπορν λέει ότι και μάλιστα να πω παρενθετικά ότι τη γραπτή δήλωση υπέγραψα μόνο οι 184 από τους 700 τόσους βουλευτές. Αυτή λοιπόν η δήλωση δείχνει ε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ αν θέλετε να απαντήσετε εκ μέρους του Συμβουλίου. Uh, concerning the regulatory environment and I think really... Ευχαριστώ. Ναι, όντως το κανονιστικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Ε, για, η και η σταθερότητα αυτών είναι πολύ σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σίγουρα το νέο πλαίσιο που προσπαθούμε να θεσμοθετήσουμε δίνει μεγάλη σημασία ε, στην νομοθετική διαδικασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε κρατικό επίπεδο, εθνικό ή ε, τοπικό επίπεδο. Ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προσφέρουν περισσότερη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε βασικούς τομείς όπως είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, όπως είναι η κατάρτιση και η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Έχουμε και άλλες, ε, άλλους συντελεστές ΦΠΑ αναλόγως με την ε, περιοχή ή αναλόγως με τον τομέα και πιστεύουμε ότι ε, έτσι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και θα δημιουργηθούν, θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει πολύ σημαντικές νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες, πρόταση αναθεώρησης της νομοθεσίας για το ΦΠΑ ώστε να αρθεί το εμπόδιο των ηλεκτρονικών τιμολογίων, της ανυπαρξίας δηλαδή αυτών. Είναι κάτι που θα μας κάνει να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα ενώ Επίσης, ε, με το σχέδιο δράσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα μειώνεται το βάρος που θα πρέπει αυτές να επομιστούν ε, και μάλιστα η μείωση αυτή θα φτάσει τα 6 δις ευρώ. Δεν μπορούν να ισχύουν τα ίδια για τις μακροεπιχειρήσεις, τα ίδια που ισχύουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει επισταμένως ε, πόσο θα βαρύνει οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές προτάσεις επιτάπητος και στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, προσπαθούμε να λύσουμε όσο δυνατόν περισσότερα προβλήματα και μάλιστα όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Τώρα, ως προς το δεύτερο ερώτημα, βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Αναφέρθηκα αυτό και στις εισαγωγικές μου ε, παρατηρήσεις. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2008 δάνεισε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1 δις ευρώ, 6% περισσότερο από ό,τι το 2007. Στόχος βεβαίως είναι να φτάσουμε σε υψηλότερα ποσοστά, να δανείζονται ε, να δανείζουμε περισσότερα χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ήμουν ακόμα μέλος αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν ήμουν υπεύθυνη για μια γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και στη δική μου γνωμοδότηση έκανα την εξή αξιολόγηση. Και πρέπει να σας το πω αυτό. ότι οφείλει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ανταποκριθεί στις ε, συνθήκες που αλλάζουν και να αλλάξει τις προτεραιότητές της, πράγμα και το οποίο έπραξε και μάλιστα τάχιστα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Σίγουρα κάποια χρήματα δεν φτάνουν στους αποδέκτες. Και ε, σε αυτό ενδεχομένως ευθύνονται ε, οι ομόλογοι, τα θεσμικά όργανα που είναι αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο εκάστοτε κράτος μέλος. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο έχει διατυπωθεί το δεύτερο ερώτημα. Είναι πολύ σημαντικό κοινοτικά χρήματα και χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να φτάσουν στους πραγματικούς τους αποδέκτες που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο βέβαια δεν μπορεί να εκφράσει επισήμως άποψη για την ε, ε, ε, δήλωση αυτή του κυρίου Κάσινγκς. Επιτρέψτε μου να περιοριστώ σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Καλώς. Πάμε στο τρίτο ερώτημα του κυρίου Παπανικολάου. Πρωτοβουλίες σε θέματα διαχείρισης υδάτων και ποσίμου νερού. Να σας πω ότι θα συνεδριάσουμε για 15 ε, λεπτά περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί λόγω του ότι καθυστερήσαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Ε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ε, παρακαλώ κύριε κύριε για το ερώτημα του κυρίου Παπα-Νικολάου. Σε απάντηση της ερώτησης του κυρίου Παπα-Νικολάου για τη διαχείριση των υδάτων θα ήθελα να σας πω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Προεδρία, για την Τρόικα μάλιστα, της, την τριμερή Προεδρία ε, Ισπανίας ε, ε, Ουγγαρίας και Πολωνίας και ε, έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την εργασία την οποία έχουν ξεκινήσει η ε, Ισπανία και το Βέλγιο και ελπίζουμε ότι θα ευωδώσει το έργο αυτό διότι το 2011 ελπίζουμε στα, να υιοθετηθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την πολιτική σχετικά με τους την πόρους που θα επικεντρωθούν σε τρία βασικά θέματα. Τα ακραία φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, λειψιδρία και άτακτη κατανομή των βροχοπτώσεων το δεύτερο θέμα είναι ο ρόλος των ε, οικολογικών ε, υπηρεσιών, ένα βασικό θέμα στο οποίο δεν αποδίδουμε αρκετή σημασία, θεωρούμε σαν δεδομένο το νερό ε, και δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι πρέπει να υπάρξουν οικολογικές υπηρεσίες για το νερό. Και το τρίτο θέμα που θέλουμε να διερευνήσουμε είναι η συνεργασία για τη διαχείριση του ίδα ύδατος και ε, διεθνώς και εντός των ε, κρατών μελών. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο ε, θα μπορέσει να δεχθεί την ανακοίνωση της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το, που θα εκδοθεί το 2011 σχετικά με τους υδάτινους πόρους, με την πρόληψη έλλειψης ύδατος στα κράτη μέλη και τέλος η Προεδρία οργανώνει ορισμένα γεγονότα, διεκδηλώσεις, ε, συνέδρια, ε, θα υπάρξουν συζητήσεις ε, για την διαχείριση πόσιμου ύδατος στην Ευρώπη και θα συζητηθεί το θέμα αυτό 21 με 25 Μαρτίου από τους αρμόδιους ε, ε, Ευρωπαίους Υπουργούς θέλουμε να ε, αναπτύξουμε και μία στρατηγική για τον Δούναβη και στα πλαίσια αυτά να βελτιώσουμε τη διαχείριση των υδατίνων πόρων. Ευχαριστώ. Ίσως αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση αλλά υπάρχουν επιπρόσθετες ερωτήσεις πρώτα από τον κύριο Παπανικό μετά από την κυρία Τικάου και μετά τον κύριο Ρούμπικ. Συμπληρώνοντας, υπενθυμίζω ότι η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 με ανακοίνωσή της και με τίτλο «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» επεσήμανε ότι θεωρεί πιθανό να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους στη δημιουργία πρόσθετων υποδομών υδροδότησης θυμίζω εξάλλου ότι πολλές απομονωμένες περιοχές στην ευρώπη ιδίως μικρές νησιωτικές ζώνες στο νότο όπως για παράδειγμα στα νησιά του αιγαίου πελάγους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης και πόσιμου νερού την ίδια στιγμή που μέθοδοι όπως η αφαλάτωση είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. το ερώτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό. Ωστόσο, δεν έχουν απαντηθεί από την άλλη. Η Ουγγρική Προεδρία θα προωθήσει συμπεράσματα του Συμβουλίου ως προς το θέμα αυτό και θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα ακραία καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε ακραία έκφραση των υδάτινων πόρων και θα έχουμε κάποια βασικά σχέδια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι και το 2012. Ο κ. Παπα-Νικολάου αναφέρθηκε στα νησιά του Αιγαίου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αυτών των νησιών. Πράγματι, αυτό ισχύει και αλλού. Οι κάτοικοι της Βαρκελόνης και της Νότιας Ιταλίας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτού του είδους τα προβλήματα. Το γεγονός δηλαδή ότι ε, μαζεύουν το νερό ε, σε δεξαμενές για να το έχουν όταν υπάρχει εξηρασία. Εμείς περιμένουμε με πολύ μεγάλη προσδοκία αγωνία τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι θα εμπνεύσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί ικανοποιητικά, ώστε όταν συζητηθεί το πολιετές χρηματοοικονομικό πλαίσιο να δοθεί η επαρκής έμφαση στους φυσικούς πόρους και κυρίως στους υδάτινους πόρους. Τώρα, ως προς τα ερωτήματα των άλλων δύο μιλητών, κυρίων Τίκα και Ρούμπικ, για το Δούναβι, θα ήθελα να σας πω ότι με μεγάλη χαρά παρακολουθήσαμε τον ε, κύριο Χάν να ε, κάνει μια εισαγωγή του σχεδίου δράσης για την ε, περιοχή του Δούναβη με ορίζοντα το 2013. Καλύπτεται σε αυτό το σχέδιο δράσης και η ξηρασία και η ποιότητα των υδάτων. Ωστόσο, ζητήθηκε από δύο κράτη-μέλη να ηγηθούν σε αυτή την προσπάθεια εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Η στρατηγική για το Δούναβι είναι μια στρατηγική που περιλαμβάνει οκτώ κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων τα έξι δεν είναι οκτώ κράτη, μεταξύ των οποίων τα έξι δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε επιπρόσθετους πόρους, μπορούμε όμως να προσαρμόσουμε τα σχέδια που δρομολογούνται αυτή τη στιγμή, να τα αλλάξουμε και να τα τροποποιήσουμε ώστε να αξιοποιούνται πιο αποτελεσματικά οι διαθέσιμοι δεν μπορεί ένα κράτος να λειτουργήσει από μόνο του από τη στιγμή που ένας ποταμό περνάει από όλε αυτές τις χώρες και τι συνδέει. Θα πρέπει να συνεργαστούμε. Κάποια σχέδια δεν θα προλάβουμε να τα εφαρμόσουμε κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας, τη Ουγγρική. Ε, η φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε το αναρκτήριο λάκτισμα το έχουμε ήδη κάνει σε επίπεδο ομάδων εργασίας αλλά και σε επίπεδο ε, Συμβουλίου Υπουργών. Ελπίζουμε στο Συμβούλιο ε, Υπουργών Γενικών Υποθέσεων θα υιοθετηθούν τα συμπεράσματα και στη συνέχεια ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση των υδάτινων πόρων και την επεξεργασία των λιμάτων. Ευχαριστώ. Εγώ θα πάω άλλη μια ερώτηση. Γιατί η κυρία ούτε είναι πολύ πιστή στην ώρα των ερωτήσεων και θα ακούσουμε και μια συμπληρωματική ερώτηση. Πρόεδρε, είμαι ευτυχής που έχουμε ακόμα το χρόνο να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή η Σύμβαση μάλλον των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι και ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση των ε, δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και η κοινότητα και τα κρατημέλη το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Θα θέλαμε να πιστήσουμε την προσοχή της ε, κυρία Βουλευτού ότι, ε, για το ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ατόμων με ειδικέ ανάγκε και θέλουμε να παρέχουμε τις προϋποθέσεις για ίση συμμετοχή στην κοινωνία των ανθρώπων αυτών, τότε θα πρέπει να εμπλακούμε στην λήψη αποφάσεων. Το Συμβούλιο το 2008 και το 2010 στα ψηφίσματά του, στις αποφάσεις τους, διαρκώς καλούσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναζητήσουν τη συμμετοχή, των, την εμπλοκή μάλλον των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες όταν αποφασίζουν για συγκεκριμένες πολιτικές. Το Συμβούλιο επίσης υιοθέτησε μια οδηγία που απαγορεύει την διακρίση επί τη βάση ε, αναπηρίας στον χώρο εργασίας. Ε, Επίση προβλέπεται η συμμετοχή των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε στι ενώσει εργαζομένων και εργοδοτών, ώστε να είναι και πραγματική συμμετοχή των ανθρώπων αυτών. Η Κομισιόν έχει μια νέα στατικική για τι αναπηρίε που υιοθετήθηκε με το περασμένο φθινόπωρο και που βασικά είναι μια απόπειρα για εφαρμογή της ε, σύμβασης του ΟΗΕ η Ουγγρική Προεδρία εξετάζει τα συμπεράσματα που θα καταθέσει για το Συμβούλιο και ελπίζουμε πως τα συμπεράσματα αυτά θα υιοθετηθούν τον Ιούνιο στην ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου. Όσον αφορά τη δημιουργία μιας επιτροπής περί δεν έχει γίνει τέτοια πρόταση στο Συμβούλιο. Να σα θυμίσω ότι το Συμβούλιο μπορεί μόνο να ασχοληθεί με προτάσει που έχουν υποβληθεί από την Κομισιόν. Αν και ε, πάντοτε εμείς ε, λαμβάνουμε υπόψη και τις απόψεις του Κοινοβουλίου, πάντως ο κανόνας είναι έτσι. Η κυρία Μπλίνκεβιτσούτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω μία επιπλέον ερώτηση επί του ιδίου θέματος. Ε, φέτος το Φόρουμ ε, Αναπηριών οργάνωσε μία συνάντηση και η Επίτροπος Ρέντιν κατά τη συνάντηση αυτή είπε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή συνθήκη για την καταπολέμηση των διακρίσεων και ε, αυτό είναι ένα σημαντικό νομοθέτημα ε, υπέρ των ατόμων με αναπηρίες. Οπότε ε, ήθελα να, γίνει, να ρωτήσω αν πρόκειται να γίνει μια αναθεώρηση αυτής της οδηγίας και αν πρόκειται τελικώς να υιοθετηθεί σχετική οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την απάντησή σας. Ε, θα προτρέψω το Συμβούλιο να ε, ε, δώσει την δέουσα προσοχή στη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία διότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι εμείς είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών. Θέλω να συγχαρώ την Προεδρία για το γεγονός ότι ε, υπάρχει μια καλή προοπτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ελπίζω να συνεχίσετε επί της ιδίας κατευθύνσεως για το μέλλον επίσης. Έχω σχετικά με τις συμπληρωματικές ερωτήσεις. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση της κυρίας Μπλινκεβιτσούτε αναφέρεται εις την ε, ε, οδηγία ενάντια στις ε, διακρίσεις. Θα μπορούσα βέβαια να σας πω ότι βεβαίως θα το επιλύσουμε διότι τέτοιες προτάσεις και τέτοιες δεσμεύσεις είναι εύκολες αλλά έχετε ε, ιδία πήραν για το πόσο δύσκολη είναι, ε, έχει υπάρξει η ε, νομοθετική διαδικασία για αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση οπότε θα επικεντρωθούμε εις την πτυχή αρχή ε, της οδηγίας που αναφέρεται στις αναπηρίες και σκοπεύουμε να κάνουμε δύο συνεδριάσεις επ' αυτού του θέματος ελπίζοντας τουλάχιστον να μπορέσουμε κάπως να προχωρήσουμε επί του θέματος. Δεν προσπαθούμε δηλαδή να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε όλο το θέμα αλλά μόνο ε, το θέμα των αναπηριών. Θα είναι όμως πολύ δύσκολο εγχείρημα διότι τα κράτη-μέλη αναφέρουν και επικαλούνται οικονομικές δυσκολίες ακόμη και στη δικιά μου χώρα, στη δικιά μου πατρίδα όπου δεν μπορέσαμε μέχρι στιγμής ε, να εφαρμόσουμε ε, τα μέτρα και να υπάρξει προσβασιμότητα για τα άτομα ε, με ειδικέ ανάγκες αλλά θα προωθήσουμε το θέμα και όπως λέγεται δεν είναι μόνο θέμα των αναπήρων αλλά και για τις νεαρές μητέρες και για άτομα τα οποία συνήθως δεν θεωρούνται σαν άτομα με ειδικέ ανάγκες. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Κόσα, πώς μπορούμε να εμπλακούμε πιο θετικά σε αυτή τη διαδικασία, ο υπεύθυνο της ομάδος για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες θα έχει προφανώς πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο με την Προεδρία και το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν δει σε πολλές περιπτώσεις ότι όταν προπορεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αισθάνονται υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τη γραμμή που διαγράφει το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει αντικείμενο προτάσεως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα διότι για την στρατηγική για τους Ρωμά αφού εσείς ψηφίσατε την σχετική έκθεση. Ελπίζουμε ότι τώρα η έκθεση αυτή θα αντικατοπτριστεί και στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τις ερωτήσεις που δεν είχαμε το χρόνο να απαντήσουμε θα τα απαντήσω γρα, γραπτός. Κύριε Χουντή, συμπληρωματική για αυτή την ερώτηση. Να συζητηθεί η ερώτηση την οποία έχω υποβάλει εκτιμώ την προσπάθεια που κάνετε και δεν θέλω να ανατραπεί η σειρά. μόνο μία παρατήρηση που δεν αφορά τον πρόεδρο συγκεκριμένα ναι παρακαλώ σύντομα θα είμαι ναι παρακαλώ δεν σας αφορά δεν είναι ευθύγη σας. θέλω να σας πω ότι επειδή έχουμε πρόβλημα με το ζήτημα του κοινοβουλευτικού ελέγχου το γνωρίζετε εσεί πολύ καλά ήταν τρει φορέ που σε ολομέλεια δεν είχαμε ερωτήσει προ το συμβούλιο και οι διαδικασίε στο τέλο καταλήγουν να συρρυκνώνεται ο χρόνο. Σα παρακαλώ λοιπόν συζητήστε στο Προεδρείο να περιφρουρείται αυτό ο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που κάνατε. Δεν θέλω να υπερβούμε το χρόνο ούτε να συζητηθεί η δική μου ερώτηση και ευχαριστώ και την Υπουργό που ήταν έτοιμη. Ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε για αυτή την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ κύριε Χούντι. Υποστηρίζω τα όσα είπατε, τα καταλαβαίνω. Δεν λαμβάνει το Προεδρείο τις αποφάσεις για το χρόνο, τη διάρκεια των συζητήσεων. η διάσκεψη των Προέδρων και προσπαθούν πάντα να βάλουν πολλά στην ημερήσια διάταξη και μετά τα μέλη του Προεδρείου ε, πρέπει να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Εγώ ζητώ συγγνώμη από όλους όσους δεν πήραν το λόγο και όπως είπε σωστά η Υπουργός θα απαντήσει γραπτό